ασυλίας σε σχέση με μια δικαστική υπόθεση στην Αγγλία και η τελευταία ανακοίνωση, η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ανακοίνωσε στον πρόεδρο πως ο κύριος Ρενάτο Σόρου φεύγει από την ομάδα αυτή και η απόφαση αυτή